Please take your seats. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. συνδιοργανώνουμε τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης. Παρευρίσκονται επίσης μέλη από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ασφαλείας και Άμυνας. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα εργαστούμε μαζί σήμερα και προσβλέπω με ανυπομονησία στη σημερινή μα συζήτηση. Δεν, δεν έχουν γίνει προτάσεις για τροποποίηση του σχεδίου ημερησία διατάξεως, οπότε μπορούμε να το εγκρίνουμε και περνούμε απευθείας στο σημείο 2 σήμερα. Μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε με την κυρία Μισελ Μπασελέ που είναι αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ και επικεφαλής εκτελεστική διευθύντρια της μονάδας ε, του ΟΗΕ για τις γυναίκες. Σας καλωσορίζουμε κυρία Μπασελέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη σημερινή μας συνεδρίαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας ε, η κυρία Μπασελέ τη συνδέσατε εξάλλου με την πρώτη σας επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να σας θυμίσω ε, διαδραματίζει πάρα πολύ ενεργό ρόλο, διαδραμάτισε μάλλον πολύ ενεργό ρόλο για τη σύσταση της ειδική υπηρεσίας για την ισότητα των φίλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στον ΟΗΕ, ούτω ώστε να συντονίσουμε τη δράση μας, να θεσπίσουμε επιχειρησιακά μέτρα, με τρόπο ώστε τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα η υπηρεσία για τις ε, γυναίκες θα έχει τους απαιτούμενους ε, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να λειτουργήσει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τεθήκατε επικεφαλής ε, με την ιδιότητά σας της αναπληρώτριας Γενικού Γενικής Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα πλέον έχει συσταθεί αυτή η ειδική υπηρεσία και περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε την παρουσίαση του προγράμματός σας και των προτάσεων σας για το μέλλον. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you very much, Madam President. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Εύα Μπριτ κυρία Εύα Ζολή, κυρία Αλεξάνδρε Γκράφ Λάνστορφ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι ευτυχής που έχω αυτή την ευκαιρία να σας απευθύνω για πρώτη φορά το λόγο ως ε, πρώτη διευθύντρια αυτής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και την ε, ενίσχυση των γυναικών, UN Women ε, με συντομία. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και προσβλέπω στην σημερινή μας συνομιλία. Η Έλενορ Ρούσβελ πριν από 60 χρόνια όταν έγινε η δήλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησε έναν κόσμο όπου τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών και η κοινωνική τους προστασία θα ήταν εγγυημένα. Ε, ζήτησε να υπάρξουν οι απαραίτητες ευκαιρίες για τη στέγαση, για την παιδεία, για την πρόσβαση στην υγεία, για την πρόσβαση στην πρόνοια, στην αξιοπρέπεια και στο σεβασμό. Μετά από 60 χρόνια και πάνω Ακόμα πόρο απέχουμε από την επίτευξη αυτών των στόχων. Όχι μόνο οι άνδρες, αλλά και εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες ολόκληρο τον κόσμο ζουν στη φτώχεια και βρίσκονται πολύ πίσω. Πάνω από το ίμιση της ανθρωπότητας υποφέρει από ανισότητες. Όταν λοιπόν ε, τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτή τη νέα υπηρεσία, ήταν σαφέ ότι ακόμα και αν έχει υπάρξει πρόοδο, οι γυναίκε και τα κορίτσια δεν είχαν τι ευκαιρίε που του αξίζουν. Όταν ε, εξετάζουμε λοιπόν ε, με την υπηρεσία μας τις γυναίκες, οι φιλοδοξίες μας είναι να έχουν τις ίδιες δυνατότητες οι γυναίκες και με την αρχή, η αρχή μάλλον της ισότητας των φύλων να είναι ενσωματωμένη σε όλες τις άλλες πολιτικές και ατζέντες. Εγώ προέρχομαι από το Παρίσι, όπου χρησιμοποιούσα την άλλη μου ιδιότητα, δηλαδή ότι είμαι πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδας ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας για την Κοινωνική Πρόνοια και εξετάζουμε μέσα στην ατζέντα G των G20 όχι μόνο οικονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές αλλά και πολιτικές που επηρεάζουν τον κόσμο, την πραγματική οικονομία και γι' αυτό ελπίζουμε ότι μέσα από το G20 θα αναπτυχθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για να υποστηριχτούν ε, τα κοινωνικά ζητήματα, γιατί είδαμε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά την κρίση όλες οι χώρες που θέσπισαν προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας όχι μόνο μπόρεσαν να αποφύγουν την κοινωνική κατάρρευση της οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά μπόρεσαν να ανταποκριθούν πολύ ευκολότερα και καλύτερα στην κρίση. Και όλα αυτά τα αναφέρω γιατί οι γυναίκε και η κοινωνική προστασία είναι αλληλένδετες. Οι γυναίκε, σε όλε αυτές τις χώρες όπως η Βραζιλία, το Μαξικό, η Ινδονησία, η Ινδία, η Χιλή, όπου αναπτύσσουμε τέτοιου είδους προγράμματα, οι γυναίκε ήταν οι βασικοί ε, παράγοντε και φορεί. Ακόμα και οι γυναίκε που είπα ότι έχουν μείνει πίσω και που είναι θύματα τόσων ανισοτήτων και διαφορών, ακόμα και βία. Εξακολουθώ να πιστεύω πως οι γυναίκες είναι οι φορείς της ανάπτυξης και της αλλαγής και της ειρήνης. Όταν μιλάμε λοιπόν για κοινωνική προστασία ή όταν μιλάμε για γυναίκες, μιλάμε για προστασία, για πρόληψη, αλλά και για ε, ενδυνάμωση των γυναικών, δηλαδή απελευθέρωση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων που έχουν οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι βέβαιη ότι οι γυναίκες μπορούν να αποτελέσουν τον καταλήτη για την αλλαγή, να προσφέρουν ε, νέα ενέργεια ε, και να φέρουν κοντά τις γυναίκες και τους άνδρες από διάφορες ε, χώρες, κοινωνίες, ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε μία πεποίθηση ότι η ισότητα των φύλων και η ισοβασμός των δικαιωμάτων της ε, γυναίκας θα είναι δυνατός μόνο αν υπάρξει πραγματική χειραφέτηση των γυναικών. Το βασικό μας θέμα λοιπόν είναι η χειραφέτηση. Όταν εξετάζουμε λοιπόν τις προτεραιότητες, αυτές ενδέονται με την ε, συνείδηση του ότι ε, πρέπει να χειραφετηθούν οι πιο αδύναμες, ε, δηλαδή συνήθως είναι οι γυναίκες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι και τα αγόρια και οι άνδρες. Πολύ συχνά θεωρούμε πως μια προτεραιότητα είναι η συμμετοχή των γυναικών και η δυνατότητα να έχουν φωνή οι γυναίκες σε όλους τους τομείς όπου οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Η έλλειψη ε, εξουσίας πολλές φορές είναι το αίτιο της ανισότητας και της απόστασης από τα τεκτενόμενα. Θα επανέλθω αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ότι είμαι πολύ ε, βέβαιη ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ ίσα δικαιώματα αν δεν υπάρχει οικονομική ασφάλεια και οικονομική αυτονομία των γυναικών. Γι' αυτό και η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών είναι εξίσου σημαντική με την πολιτική χειραφέτηση του. Τρίτη προτεραιότητα είναι να σταματήσει αυτό το φοβερό δράμα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και είναι μια παγκόσμια πανδημία και εδώ στην Ευρώπη. Τέταρτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της εφαρμογής της ατζέντα ε, των γυναικών για την ειρήνη και την ασφάλεια και τέλος εξασφάλιση της ισότητας, ε, της προτεραιότητας μάλλον, της ισότητας των φύλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε όλες τις στρατηγικές και τις πολιτικές. Να πω δύο λόγια παραπάνω για αυτές τις, ε, τους βασικούς Καταρχήν ανέφερα την ε, χειραφέτηση των γυναικών, τη συμμετοχή και την ε, ηγετική ικανότητα των γυναικών. Και εσείς εδώ είστε πολλοί άνδρες και γυναίκες που μπορείτε να αποδείξετε πως είναι δυνατό κάτι τέτοιο γιατί δράτε σαν μέντορες, σαν πρότυπα και μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι γυναίκες μπορούν να κρατήσουν σημαντικές θέσεις σε πόστα λήψης αποφάσεων. Ε, μόλις επισκέφθηκα το Καϊρό και μάλιστα ορισμένου από εσάς σας είδα και εκεί ως τμήμα της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ, ως μέρος μάλλον της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ και θέλω να σας πω πόσο με χαροποίησε που είδα γυναίκες νέες και λιγότερο νέες αποφασισμένες να εξακολουθήσουν να παίρνουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ώστε να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Και ήθελα να τονίσω τον ρόλο κλειδί που έπαιξαν οι γυναίκες για τις αλλαγές σε ολόκληρη την περιοχή και ελπίζω πως αυτό θα αντικατοπτριστεί και στις θεσμικές αλλαγές που τώρα συζητώνται, γιατί πιστεύω πως οι γυναίκες θα πρέπει να είναι στην καρδιά αυτών των συζητήσεων, όπως ε, ήταν στην καρδιά της πλατείας ε, Ταχρή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν δύο σημαντικές προκλήσεις. Ε, κάτι που είναι ιδιαίτερα προσφυλές σε μένα, γιατί και στη Χιλή ζήσαμε μια τέτοια διαδικασία, είναι η μετάβαση στη δημοκρατία. Και η μετάβαση στη δημοκρατία σημαίνει πολλές ε, νομικές αλλαγές, ενίσχυση των πολιτικών οργανώσεων, ανάπτυξη εκλογικής νομοθεσίας, εξασφάλιση της ε, ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας έκφρασης. Αλλά η δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο εκλογή ελεύθερη, είναι κυρίως η εγγύηση του πλουραλισμού και της ένταξης. Οι γυναίκες δηλαδή που ήταν εκεί να μπορέσουν να παίξουν ρόλο στον ανασχηματισμό της κοινωνίας τους. Το άλλο όμως σημαντικό πράγμα, γιατί η δημοκρατία είναι ναι, χειραφέτηση, αλλά κάτι ακόμα σημαντικό, είναι ότι ε, ε, η δημοκρατία σημαίνει και κοινωνική δικαιοσύνη ή κοινωνική πρόνοια. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η δημοκρατία πρέπει να αποδώσει καρπούς. Γιατί η φτώχεια είναι πολύ μεγάλη, υπάρχουν το πάρα πολύ αναλφάβητοι, υπάρχει πολύ ψηλός ε, πληθωρισμός, μεγάλο ποσοστό ε, ανέργων νέων και πιστεύω και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα ότι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική πρέπει να τα στηρίξουμε σοβαρά γιατί διαφορετικά οι λαοί θα απογοητευθούν. Εξάλλου, ε, είναι γνωστό ότι όταν βρέχει στην Αίγυπτο, ο υπόλοιπος αραβικός κόσμος ανοίγει τις ομπρέλες του. Δηλαδή θεωρούν την Αίγυπτο ως πρότυπο για οτιδήποτε γίνεται στον αραβικό κόσμο. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Μιλάμε τώρα για ισότητα των φύλων. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η πρόοδος στην ισότητα των ε, φίλων απαιτεί αλλαγή και του status quo. Αναγνωρίστηκε αυτό στην πλατφόρμα του Πεκίνου. Οι, τα, οι πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών υποστηρίχτηκαν από τη διεθνή κοινότητα ώστε να αναλυφθούν θετικέ δράσει για να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα γυναικών ηγετών και να προωθηθεί η θέση της γυναίκας. Αν δούμε όμως τον κόσμο σήμερα, η μικρότερη πρόοδος για τις γυναίκες είναι στο πολιτικό επίπεδο. Έχουμε μέσο όρο 19% γυναικών βουλευτών και αυτός είναι ένας μέσος όρος που προέρχεται από το μεγαλύτερο ποσοστό στον κόσμο που είναι στη Ρουάντα, όπου έχουν περίπου 54,7%. Και <coughs> είναι πολύ σημαντικό το Νεπάλ με 34% ποσοστό γυναικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην περιοχή του Νοτίου Ειρηνικού. Έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά είναι πολύ αργή. Τον Ιανουάριο του 2011, αν δούμε τους στόχους του Πεκίνου που ετέθησαν πριν από 15 χρόνια, θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα του 30% ε, γυναικείας εκπροσώπησης στα κοινοβούλια και μόνο 28 χώρες το έχουν πετύχει αυτό το στόχο συμπεριλαμβανομένων 7 στην, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. 28 χώρες ε, σε ένα μεγάλο φάσμα οικονομικής ανάπτυξης δίνουν, δείχνει ότι η πολιτική συμμετοχή μπορεί να υπάρξει μέσω της δέσμευσης της εφοσίωσης των ίδιων των πολιτικών ηγετών. Μόνο πέντε χώρες δεν χρειάστηκαν ειδικού μηχανισμούς για την πρόθεση των γυναικών. Οι υπόλοιπε 23 χρειάστηκε να υιοθετήσουν κάποια μορφή ποσόστοσης ή θετικής δράσης, ή μέτρων μάλλον θετικής δράσης, για να μπορέσουν να φτάσουν το ποσοστό του 30%. Όσον αφορά λοιπόν την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ε, σε όλα τα πολιτικά επίπεδα, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης, ε, ε, κατάρτιση, για να μπορέσουν να φτάσουν σε πολιτικές θέσεις και να μπορέσουν να κάνουν σωστές πολιτικές εκστρατείες. Αυτό θα σημαίνει και οικονομική χειραφέτηση. Πριν από 8 χρόνια η Νορβηγία θέσπισε ένα, μια νομοθεσία υπέρ των γυναικών. Σήμερα οι γυναίκες καλύπτουν το 32% των ε, θέσεων λήψης αποφάσεων ε, στην Νορβηγία. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία ε, έχουν ε, υιοθετήσει παρόμοια νομοθεσία. Μέχρι το 2015 πρέπει να έχει επιτευχθεί παρόμοιο στόχο. Το ίδιο και στην Ιταλία και στην ε, Γαλλία. Και αυτό έχει νόημα ότι, γιατί το ταλέντο είναι πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα, αλλά το γυναικείο ταλέντο δεν χρησιμοποιείται πλήρω. Στην Ευρώπη οι γυναίκε αποτελούν το 45% του εργατικού δυναμικού. Όμω μόνο το 11% των υψηλά ειστάμενων στελεχών των επιχειρήσεων οι μελέτε δείχνουν ότι όταν αυξηθεί ο αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, η οικονομική απόδοση βελτιώνεται. Η υπηρεσία μας συνεργάζεται με την ε, υπηρεσία Global Compact για να υποστηρίξει τις αρχές και να προωθήσει τις αρχές χειραφέτησης των γυναικών. Και αυτές οι αρχές καλούν τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θα αντιπροσωπεύουν το 30% των ομάδων που είναι για, υπεύθυνες για την λήψη αποφάσεων και θα λαμβάνουν ισότιμους μισθούς για ισότιμες θέσεις. Η διαφορά ε, στη μισθοδοσία ε, φτάνει το 80% ε, με τους άνδρες. Θέλω να ε, βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και να υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Επίσης, θέλω να συνεργαστούμε με ε, πολυμερεί εταίρους και κυβερνήσει για να ε, εξασφαλιστεί πλήρω η οικονομική ασφάλεια των γυναικών και τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της ε, αξιοπρεπού εργασία και τη κοινωνική προστασία. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία σε ένα κόσμο σταθή και στι τιμές των τροφίμων και στι τιμέ των εμπορευμάτων και σε άλλους τομείς που πλήττονται οι γυναίκε. Στι πιο φτωχέ χώρες και στι πιο ευάλωτε χώρες η ενδυνάμωση των γυναικών, η ενίσχυση των γυναικών είναι κλειδί για μα. Ε, στις 8 Μαρτίου ήμουν στη Λιβερία και πολλέ γυναίκε έχουν ε, την οικονομία στα χέρια τους, εργάζονται σε αγορές, έχουν ε, ε, αγροκτήματα, ε, εμπορικά καταστήματα. Εκεί θέλουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες των γυναικών, να τους μάθουμε να διαβάζουν. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή κανείς ηλικιωμένες γυναίκες να μαθαίνουν ε, ανάγνωση, να καταπολέμει τον ε, αναλφαβητισμό και μου έδειξε ότι πώς μπορεί να διαβάζει και μπορεί να διαβάζει και τα ψηλά γράμματα και μου είπε κανείς δεν θα με κοροδέψει πια γιατί ξαναδιαβάζω. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό και επίσης οι γυναίκες είναι παραγωγή, παράγουν πάρα πολλά προϊόντα και ε, τους μαθαίνουμε πώς ε, να προσθέτουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους, να έχουν πρόσβαση σε αποθήκες, σε εμπόριο, ε, να μπορούν να τα αποθηκεύουν για να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές. Αλλιώς είναι καταδικασμένες να παραμένουν στη φτώχεια για το υπόλοιπο της ζωής τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Αλλά και στον αναπτυγμένο κόσμο και στην ε, Ευρώπη, παρόλο που οι γυναίκε είναι σε πολύ καλύτερη θέση, απομένουν πάρα πολλά για τι μετανάστριε, για τι εργάτριε, για τι ε, εργαζόμενε κατοίκων κτλ. Και έρχομαι τώρα στην τρίτη θεματική ε, ενότητα που είναι η πάταξη της βίας κατά των γυναικών παγκοσμίως. Είναι πραγματική πανδημία. Γνωρίζουμε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό παντού, σε όλο τον κόσμο και για τις γυναίκες Και γνωρίζω ότι είναι και προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό το θέμα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση και τους νόμους που αυξάνονται για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ε, παραμένει μάστιγα και ε, επιδημία, πανδημία σε όλο τον κόσμο. Ε, είναι πάνω από 100 οι χώρες που έχουν νομοθεσία, αλλά δεν την εφαρμόζουν συλλαμβάνονται οι πέτοι, αλλά οι δικαστές του αφήνουν ελεύθερου γιατί δεν το θεωρούν σημαντικό. τρία τέταρτα των γυναικών σε κάποια μέρη έχουν ε, δηλώσει ότι έχουν υποστεί σωματική ή ε, σεξουαλική βία σε κάποια στιγμή τη ζωής του. 20% των γυναικών στην Ευρώπη ε, από στενές σχέσεις ομολογούν ότι έχουν υποστεί τέτοια βία σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Γυναικών και αυτό έχει σημασία και μεγάλο κόστος για τη ζωή τους, την υγεία, την παραγωγικότητα, την επίδοση στο σχολείο, ε, το, τα δημόσια οικονομικά και σε όλες, χώρες, όλες τις χώρες, όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες. Επίσης δεν έχουμε καταφέρει να υπολογίσουμε το κόστος, όχι μόνο το ανθρώπινο κόστος, αλλά τι σημαίνει αυτό για την οικονομία ενός κράτους. Εγώ πιστεύω ότι είναι η πιο διαστραμμένη βία και η πιο διαστραμμένη παραβίαση των γυναικείων δικαιωμάτων, η βία κατά των γυναικών. Στην Ινδία έχει δείξει μια μελέτη ότι για κάθε επεισόδιο βίας χάνονται πέντε εργάσιμες ημέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από μερικά χρόνια βέβαια, 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο υπολογίζονται απώλειες το 2005. 135 δις ε, αλλού και στην Αυστρία το 2010 τους κόστισε 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα ε, που έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος και ανθρώπινο και κοινωνικό αλλά και οικονομικό και διαφορετικές ε, επιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει η μάστιγα αυτή, αλλά θα, θα πρέπει να ε, την αντιμετωπίσουμε σε πολλά μέτωπα, να υποστηρίξουμε μηχανισμούς ε, επιβολής του νόμου και να δοθεί προσοχή και στην πρόληψη και στην ε, θεραπεία και να συμμετέχουν όλοι οι τομείς κοινωνίας και βέβαια οι άνδρες και τα γόρια. Θα πρέπει εκείνοι να αισθανιστούν και να είναι οι πρωταθλητές ε, της υπόθεσης αυτής υπέρ των γυναικών και των κοριτσιών. Και τουλάχιστον οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν ε, πέσει θύματα βίας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε δικαιοσύνη για να αποφευχθεί η επανάληψη της κατάχρησης. Τους επόμενους μήνες θα συνεργαστώ ε, στενά με κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών προς τον σκοπό αυτό. Και με τη UNICEF. Στο παρελθόν υπήρχαν ασφαλείς πόλεις ε, ονομαζόμενες safe cities για ε, τα κορίτσια και τις γυναίκες. Χρειάζεται συνέχιση αυτής της προσπάθειας από κοινού για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια καταφύγια για τις γυναίκες και τα κορίτσια αυτά. Την περασμένη εβδομάδα ξέρω ότι ε, εγκρίνεται μια έκθεση της Προέδρου κυρίας Φένσον για ένα πλαίσιο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών για να αναγνωριστεί ε, η ε, σεξουαλική βία και ο βιασμός εντός του γάμου ως αδίκημα και να βοηθηθούν και οι οικογένειες και οι γυναίκες να ξεπεράσουν τα τραύματά τους αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε τα πιο φρικτά ε, εγκλήματα και σεξουαλικά και ε, εγκλήματα φύλου συμβαίνουν σε περιοχές σειράξεων ή μετά τη σύραξη. Οι φωνές τους δεν ακούγονται το γυναικό όμως αυτών στις ε, νευτικές διαπραγματεύσεις. Η UN Women διαπίστωσε ότι σε 24 ειρηνευτικές διαδικασίες των τελευταίων 20 ετών οι γυναίκες είναι λιγότερο από 8% των διαπραγματευτικών ομάδων. Αλλά πάνω από 500 συνευτικές συμφωνίες που είχαμε μετά το ψυχρό πόλεμο, μόνο σε 16 περιπτώσεις αναφέρθηκε η λέξη γυναίκα και μόνο σε 8 αναφέρθηκε ο όρος σεξουαλική βία, η βία με βάση τον φίλο. Και σας είπα είναι πάνω από 500 οι συμφωνίες μετά ε, το ψυχρό πόλεμο και παντού οι γυναίκες ήταν θύματα και θύματα σεξουαλικής βίας και ε, αυτή η βία ήταν ε, πολεμικό όπλο. Πέρυσι γιορτάσαμε τα 10 χρόνια από το ψήφισμα 1325 του ΙΕ, αλλά η ε, πρόοδος είναι πάρα πολύ αργή. Είναι προτεραιότητα για μας αυτό το θέμα και με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία ως διαμεσολαβήτριες ε, και ε, για την πρόληψη ε, της συστηματικής σεξουαλικής βίας. Να έχουμε συστήματα έγκαιρης πρόορης ε, προειδοποίησης, να είναι εκπαιδευμένο και το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών. Καλούμε όμως ε, τις γυναίκες και τα κράτη να στέλνουν περισσότερες γυναίκες στους κιανόκρανους ή στην αστυνομία. Στη Λιβυρία είχαμε πολύ καλή εμπειρία με Ινδές αστυνομικίνες που ε, ήταν επιτόπου και οι γυναίκες ε, είχαν ε, πολύ μεγαλύτερη άνεση. Εγώ διατέλεσα και υπουργό άμυνα στη χώρα μου. Είναι σημαντικό να βλέπουμε τι γυναίκε ένστολε, ένοπλε, γιατί αυτό δείχνει ότι έχουν εξουσία και ισχύ ε, οι γυναίκε και ψυχολογικά είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον πληθυσμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη ε, που έδωσε στην εφαρμογή του ψηφίσματο 1325 και θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το να εορτάσει την επέτειο τη δέκατη επέτειο του ψηφίσματος και ε, βοηθάει ε, να εφαρμοστεί και αυτό το ψήφισμα και τα επόμενα ε, για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Και πάλι, όταν άρχισα να μιλώ, είπα ότι αν θέλουμε ισότητα φύλων, χρειάζεται να δώσουμε ισχύ στις γυναίκες, να ενδυναμωθούν οι γυναίκες παντού. Παντού. Αν γυναίκες δεν έχουν φωνή, αν οι γυναίκες δεν έχουν ισχύ, ε, δεν κάθονται ποτέ στα τραπέζια λήψη αποφάσεων. Είναι πάντα εκτός. Τι βλέπουμε στις ειρηνευτικές διαδικασίε. Ποιο διαπραγματεύεται, εκείνοι που έχουν ισχύ, εκείνοι που έχουν τα όπλα, εκείνοι που έχουν ε, την ισχύ. Το Νεπάλ είναι ενδιαφέρον να το θυμηθεί κανείς. 40% του μαοϊκού στρατού ήταν γυναίκες και αμέσως μετά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και στην νομοθεσία και στην ε, νευτική προσπάθεια. Εγώ δεν θέλω να συνηγορώ υπέρ των όπλων, αλλά όταν οι γυναίκες έχουν διατελέσει ένοπλες έχουν και άλλη διαπραγματευτική ισχύ και εξουσία. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομεί όπου ε, η υπηρεσία των ΗΠΑ για τις γυναίκες συνεργάζεται με άλλους. Ε, για τις για τα δικαιώματα των γυναικών, την υγεία των γυναικών, για την καταπολέμηση του AIDS και του HIV, για την καταπολέμηση των μητρικών θανάτων στο δοκετό, για ένα σωρό θέματα ε, τα οποία μας απασχολούν, υποστηρίζουμε τις γυναίκες, προσπαθούμε να τις ε, ενισχύσουμε. Ε, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η UNESCO Όλα αυτά είναι σημαντικοί οργανισμοί, συνεργαζόμαστε μαζί τους και ξεκινούμε προσπάθειες κτλ. Θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένες από τις προτεραιότητές μας και κέντρα βάρους και όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ φιλόδοξη η στόχη μας, αλλά χρειάζεται. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μικρή κλίμακα, πρέπει να έχουμε μεγάλα σχέδια. Και ο στόχος είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, για την ενίσχυση ε, με ε, Τη συνεργασίες με το UN Women για στρατηγική ε, πραγματικά κοινή συνεργασία και μεσοπρόθεσμη. Θέλω να συζητήσω τη συνεργασία μας, αλλά γνωρίζω πολύ καλά και ε, το τι περιμένουν από εμά, αλλά και ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πάντως θα τις αντιμετωπίσουμε. όταν τους δίνουμε την ευκαιρία δεν έχουν όρια οι δυνατότητες των γυναικών. Από τη την ε, ζωή της οικογένειας μέχρι τις πιο σκληρές συνθήκε και την πολιτική Υπουργή Οικονομικών, Εξωτερικών, ακόμα και Αρχηγή Κρατών. Πραγματικά θα πρέπει να απελευθερώσουμε την ενέργεια και τη δύναμη των γυναικών, να το συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες προς όφελος όλων. Ευχαριστώ πολύ. Ένα θερμό ευχαριστώ προς την κυρία Μπασελέ. Ήσασταν κατατοπιστικότατοι σε αυτή την πληρέστατη αρχική σας παρουσίαση. Μιλήσατε για τις ε, πολιτικές, οικονομικές ελευθερίες, την καταπολέμηση της βίας. Καλύψατε όλες τις ε, πτυχές. Σας ευχαριστούμε και πριν δώσω το λόγο ε, στον εκπρόσωπο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, θα ήθελα να σας πω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα χρόνου. Δεν θα έχουμε καθόλου χρόνο γιατί πάρα πολλοί θέλουν να μιλήσουν. Και προφανώς θέλουμε να δώσουμε και την ευκαιρία στην κυρία Μπασελέ να σχολιάσει κατόπιν τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Θα είμαι πολύ αυστηρή λοιπόν. Θα περιορίζω το χρόνο αγόρευσης. Ας ακούσουμε τώρα την Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο κύριος Λάμπστορφ θα πάρει το λόγο. Είναι πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ, ο κύριος Λάμπστορφ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε από πλευρά τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τη Ομάδα Εργασία για τις Σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Ήδη κάναμε μια συνεδρίαση, την ετήσια συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, πριν αναλάβετε το αξίωμά σα ε, και σα συγχαρήκαμε για το διορισμό σα στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας προφανώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτή την υπηρεσία του ΟΗΕ και θεωρούμε ότι η προώθηση της όταν των δύο φίλων και η προστασία και η χειραφέτηση των γυναικών είναι κέρια ζητήματα. Θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία που μας ανησυχούν όλους ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας. Πρώτον, ε, συντονισμό ε, με όλου του υπόλοιπου οργανισμού ε, του ΟΗΕ. Εμεί έχουμε ένα περίπλοκο σύστημα συντονισμού, χρονοβόρο τι περισσότερε φορέ. Δεν διαφέρουν και πολύ τα πράγματα στον ΟΗΕ. Σκέφτομαι την εντολή τη UNFPA, που φυσικά ασχολείται εντελεχώ με τα θέματα των γυναικών. Υπάρχει καλό συντονισμό. Αναφερθήκατε στη UNICEF, στη UNESCO. Θα θέλαμε να υπάρχουν συνέργειε ανάμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς εστιάζοντας τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τα δικαιώματα στον τομέα της υγείας, όλα τα δικαιώματα των γυναικών. Όλα αυτά μας απασχολούν στην Επιτροπή μας. Κάτι ακόμη πιο σημαντικό από τη δική μας ε, ε είναι το ψήφισμα 3025 για τις γυναίκες σε ένοπλες σειράξεις. 500 ειρηνευτικές συμφωνίες, αναφερθήκατε συγκεκριμένα σε 16 ειρηνευτικές συμφωνίες, και βλέπουμε την διάδοση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών στο Ανατολικό Κονγκό παραδείγματος χάρη χρησιμοποιείται ως ε, πολεμικό όπλο αλλά και σε, άλλα, ε, σε άλλες εμπόλεμες ζώνες. Η Μάργκρετ Βάλμστρομ ε, διορίστηκε ως ειδική εκπρόσωπος για τη βία σε, στις ένοπλες σειράξεις για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο που πλήττει τις ε, γυναίκες. Ε, η ειρηνευτική διαδικασία τώρα Πραγματικά το μόνο που μπορώ να κάνω να επιβεβαιώσω, να υπερθεματίσω αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ε, να στελεχώνουμε, ε, χρησιμοποίησα στα αγγλικά τον όρο MAND, είναι λάθος όρος, ε, τέλος πάντων στα ελληνικά να στελεχωθούν αστυνομικές και στρατιωτικές υπηρεσίες με γυναίκες, ούτως ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Το παράδειγμα που δώσατε είναι ένα απτό, επιτυχημένο παράδειγμα τέτοιας δράσης και θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλους να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, δηλαδή να στελεχώνουν αποκλειστικά και μόνο με γυναίκες διάφορες υπηρεσίε, ε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ επιτυχημένη αυτή η πρωτοβουλία. Σα σας ευχαριστούμε κύριε Λάμστορφ. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Εύα Ζολή, την πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είναι τιμή για μένα, ευκαιρία που έχω να καλωσορίζω την κυρία Μπασελέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξ ονόματο τη Επιτροπή Ανάπτυξη θέλω να σα πω πόσο σημαντικό θα είναι το έργο σα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση των γυναικών δεν βελτιώθηκε και ακούσαμε από το Σουδάν, ακούσαμε από το Κονγκό ε, ανθρώπους στις ακροάσεις για ε, μαζικές βιασμούς τρομακτικούς γυναικών και επίση γνωρίζουμε ότι οι φτωχότεροι των φτωχών είναι γυναίκες. Παράγουν τροφή για τον κόσμο ολόκληρο, αλλά δεν έχουν ε, πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Η δυνάμωση των γυναικών, η ε, ενίσχυση τους δεν ήταν ε, επιτυχής. Αν είδατε τι έγινε στις γαλλικές εκλογές την περασμένη Κυριακή τις τοπικές, τα κόμματα στη Γαλλία προτιμούν να πληρώνουν το πρόστιμο παρά να έχουν υποψήφιες γυναίκες. Και το βασικό κόμμα, το μεγαλύτερο, κατέβασε μόλις έξι γυναίκες. Μιλήσατε για τον νόμο στην Νορβηγία, για τις ε, γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, ότι ήταν επιτυχία. Ε, έγινε άλλος όταν προτάθηκε το νομοσχέδιο αυτό στην Νορβηγία και προτάθηκε ως εξής. Εάν δεν ε, συμμετέχουν 40% των γυναικών ε, μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 40% να απαρτίζεται από γυναίκες, τότε η εταιρεία διαλύεται. Ε, εκαθαρίζεται, δεν είναι να πληρώσει ένα πρόστιμο και να την γλιτώσει. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη υποψήφια ε, επικεφαλής ε, αυτής της υπηρεσίας του ΙΕ. Είστε η μητέρα όλων μας, από την προσωπική σας ζωή, από την ιστορία της οικογένειάς σας. Πραγματικά έχουμε εγγύηση ότι θα φροντίσετε πολύ καλά την κατάσταση των γυναικών σας. Ευχαριστώ που ήρθατε και καλή σας τύχη. Eh, σας ευχαριστούμε τώρα. Θα δώσουμε το λόγο στους ε, συντονιστές ε, της Επιτροπής Γυναικών. Η κυρία Έντιτ Μπάουερ θα πάρει πρώτη το λόγο εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας κυρία Μπάουερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ενώπιόν μας κυρία Μπασελέ και ε, ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να έχουμε μια μικρή δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Βεβαίως, κάθε περιφέρεια έχει τα προβλήματά της. Με υψηλές ή χαμηλότερες προτεραιότητες κάθε φορά αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου και εγώ να σας αναφέρω μια επιτυχία μας Μόλις προχθές το Συμβούλιο ενέκρινε και υπέγραψε νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση ε, τη διακίνηση ανθρώπων. Βέβαια, είναι λίγο πιο σύγχρονη η νομοθεσία από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, την αντίστοιχη. Πάντως, δεν πειράζει. Νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο είναι ε, επιτυχία. Κάτι άλλο όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι πριν από ένα χρόνο περίπου επισκεφτήκαμε τα Ηνωμένα Έθνη και τότε ήταν υπό προετοιμασία η νέα υπηρεσία σας. Και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηγόντων σας. Τότε συζητήσαμε πολλά θέματα και επιτρέψτε μου να σας φέρω ένα μόνο. Γιατί έχουμε χρονικό περιορισμό. Η μετρική θνησιμότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πάνω από 500.000 γυναίκες πεθαίνουν στο κετό ή κατά τη διάρκεια της σκιοφορίας, ε, από επιπλοκές της κοίησης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε πραγματική ουσιαστική επιτυχία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να χάνουμε 500.000 γυναίκες στο τοκετό ε, τη σήμερα ημέρα. Σας ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής ε, είναι η κυρία Εστρέλα. Έχετε και εσείς δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μπασελέ εξ ονόματος ε, της πολιτικής ομάδας σοσιαλιστών και δημοκρατών. Είναι τιμή για μας που ήρθατε και μπορούμε να έχουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Προφανώς χαιρόμαστε για το διορισμό σας, το είπα, το αξίωμα της Χιλής στο παρελθόν, τώρα είστε στο ΝΟΙΕ. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι προσδίδεται από το ΝΟΙΕ ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ισότητας των δύο φύλων και προφανώς υπολογίζουμε στη δική σας αφοσίωση την οποία καταδείξατε ανέκαθεν για τα ζητήματα αυτά. Αναφερθήκατε σε ένα θέμα και το τονίσατε ιδιαίτερο στο θέμα της ε, βίας ε, λόγω του φίλου. Δώσατε κάποια στατιστικά στοιχεία που αποκαλύπτουν ε, την σοβαρότητα του προβλήματος και έχει αναδειχθεί ήδη αυτό το θέμα σε προτεραιότητα από ό,τι μας είπατε. Πώς, με ποιο τρόπο, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με το, την υπηρεσία UN Women του ΟΗΕ, μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να συμβάλλουμε ώστε να μειωθεί ε, το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Κάτι άλλο, ένα ιδιαίτερα προσφυλές θέμα για μένα. Ε, όταν γίνατε πρόεδρος, σας ρώτησαν πώς θα συμφιλιώσετε την ε, οικογένεια οικογενειακή σας ζωή με τις ε, σοβαρές ευθύνες ε, του υπάτου αξιώματος. Μα γιατί το ρώτησαν σε εσάς, τους άντρες δεν το ρωτάνε ποτέ, μόνο στις γυναίκες το ρωτάνε. Πώς θα ε, συμφιλιώσετε την οικογενειακή και την επαγγελματική σας ζωή. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όταν μπαίνει στην πολιτική σκηνή η γυναίκα, αλλάζει η γυναίκα. Όταν ε, μπαίνουν πολλές γυναίκες στην πολιτική, τότε αλλάζει η πολιτική. Αυτό συνδέεται με το θέμα των ποσοστώσεων. Μπορείτε ε, να μας το εξηγήσετε γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση τότε, γιατί εξηγήσατε έτσι αυτό το φαινόμενο, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Ευστρέλα. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων τώρα θα ακούσουμε την κυρία Παβανόβα για δύο λεπτά επίσης. Παρακαλώ. Σας, Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπατσελέτο, αν διαβάζει κανείς ε, το βιογραφικό σας σημείωμα ε, βλέπω ότι οι σταδιοδρομίες μας μοιάζουν και εγώ ξεκίνησα ως παιδίατρος, ε, τώρα είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ξέρω πού θα φτάσω, αλλά πάντως εσάς συγχαρητήρια. Έχετε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και δύσκολο, γιατί όπως είπε η συνάδελφος Εντίτ Μπάουερ, είχαμε μεγάλες προσδοκίες από το στόχο της χιλιετίας και χθε εδώ στο Κοινοβούλιο Είχαμε την ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το AIDS και για τους ε, πολιτισμούς ανάπτυξη και συζητήσαμε για τους στόχους 4 και 5 του χιλιετίας και διαπιστώσαμε ότι εδώ και 11 χρόνια το 1 τρίτο έχουμε φτάσει και μας μένουν μόνο 4 χρόνια και δεν νομίζω πως θα επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Για τα παιδιά ε, συνδέεται αυτό με τη στόχο 4, αλλά νομίζω πως πάει χέρι με χέρι με τη χειραφέτηση των γυναικών, το στόχο 3. Η αικαιρεότητα των στόχων της χιλιετίας λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Σκοπεύεται να ενισχύσετε περισσότερο τις δραστηριότητε ε, της ε, υπηρεσίας για τις γυναίκες και να οθήσετε τις εργασίες προς την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Και η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τα δικαιώματα των γυναικών σε εμπόλεμες ζώνες και κυρίω τα όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Εμεί ελπίζουμε πω αυτέ οι επαναστάσει θα, θα φέρουν περισσότερα δικαιώματα για τι γυναίκε, αλλά απ' την άλλη ανησυχούμε μήπω υπάρξει, ε, ε, επικρατήσουν οι Ισλαμιστέ και ποιες θα, ποια θα ήταν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε σε συγκεκριμένες ε, περιοχέ ώστε να εγγυηθείτε τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εξ ονόματος των Πρασίνων. Στην Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Θα ακούσουμε την κυρία Κιλ Νίλσεν για 1,5 λεπτό. Κυρία Κιλ Νίλσεν, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπασιλέ που ήρθατε να μας ακούσετε. Ως εισηγήτρια για τις γυναίκες και τις κλιματικές αλλαγές για την Επιτροπή των Γυναικών παρακολουθώ την κατάσταση των γυναικών με μέγα ενδιαφέρον και η έκθεση που θα υποβάλλω θα συμπεριλαμβάνει συστάσεις για την λήψη υπόψη της των φύλων ε, και θα ήθελα να γνωρίζω την θέση της Υπηρεσίας Γυναικών του ΙΕ για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για τις κλιματικές αλλαγές και τις γυναίκες και πώς θα ληφθούν αυτές οι στάσεις υπόψη αυτού του είδους της παγκόσμιας διασκέψης. Επιπλέον, εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Διεθνή Επιτροπή Γυναικών που είναι ένα συνασπισμό Παλαιστινίων, Ισραηλινών γυναικών και διεθνών γυναικών με βάση το 1325 το ψήφισμα του ΟΗΕ και που στηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών στην επίλυση της ε, ισραηλο-παλαιστινικής κρίσης υπέρ μιας ε, βιώσιμης ειρηνικής λύσης. Όλο και περισσότερο οι Παλαιστίνες και οι Ισραηλινές γυναίκες δεσμεύονται στην μη βίαιη αντίσταση κατά της κατοχής. Την περασμένη 12η Μαρτίου ε, ε, αψήφισαν την απαγόρευση να διαδηλώσουν ε, κοντά στην Βιθλέμ. Μπορείτε, κυρία Μπασλέ, μπορείτε να με διαβεβαιώσετε για τη στήριξή σας προς αυτόν τον συνασπισμό που συγκεντρώνει διαμεσολαβήτριες για την ειρήνη. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε, κυρία Κιλ από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Ο κύριος Σιμάνσκι θα πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ εξ ονόματος ε, της ομάδας μου να καλωσορίσω την κυρία Μισελ Μπασολέ στη συνεδρίασή μας σας ε, συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Πραγματικά η κοινωνία μας χρειάζεται ανθρώπους στρατευμένους και προσιλωμένους στο έργο τους. Και η δική μου ομάδα είναι προσιλωμένη πολύ στα δικαιώματα των γυναικών. Εδώ, στην Επιτροπή Γυναικών, εκπονούμε αυτό το καιρό μία έκθεση για ε, τις γυναίκες επιχειρηματίες αλλά και για την υπέρβαση των εμποδίων και την κατάργηση των εμποδίων ε, των ε, γυναικών εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γυναίκες όμως χρειάζονται στην Ευρώπη και οικονομική υποστήριξη, εκτός από την υποστήριξη για τα δικαιώματά τους, για να συμφιλιώνουν ακριβώς τον εργασιακό με τον οικογενειακό τους βίο. Και στην πολιτική συνοχής ε, δεν θα πρέπει να δημιουργούμε μόνο θέσεις απασχόλησης, αλλά να φροντίζουμε οι θέσεις αυτές να είναι βιώσιμες, αηφόρες και με σωστή αμοιβή. Επίσης γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα των φτωχών εργαζομένων είναι φτωχές εργαζόμενες. Και ε, χρειάζεται ενίσχυση λοιπόν των γυναικών και στον κοινωνικό τομέα. Παραμένει μεγάλη διαφορά και στην αμοιβή ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστούμε από πλευράς ε, της GUNGL, ε, η κυρία Φιγκυρέιντο θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε, με τη σειρά μας. Θα θέλαμε να χαιρετήσουμε την κυρία Μπασλέ, να την ευχαριστήσουμε για το, την επιτέλεση των καθηκόντων της. Πέρσι ένα κλιμάκι της ομάδας GUNGL ε, μετέβη στον ΟΗΕ και συζητήσαμε αυτό το θέμα. Προφανέστατα τότε συμφωνήσαμε ότι ο στόχος είναι να προβληθούν τα βασικά και σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η διακριτική μεταχείριση, το γυναικείο πρόσωπο της ένδυας γενικότερα στον κόσμο, όχι μόνο στις φτωχότερες χώρες, όχι μόνο στις ε, χώρες ε, όπου υπάρχουν ένοπλες σειράξεις, πόλεμοι, και τα μεγαλύτερα θύματα πάντοτε είναι οι γυναίκες. Αλλά αυτό ισχύει και σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Εξακολουθούν να υπάρχουν ε, ε, φαινόμενα διακριτικής μεταχείρισης, εμπορίας ανθρώπων, πορνεία. Και σε αυτά θα πρέπει να αποδώσουμε την δέουσα προσοχή, διότι ε, εκατομμύρια γυναίκες ετησίως πέφτουν ε, θύματα ε, τέτοιων ε, κυκλωμάτων πορνείας και εμπορίας ανθρώπων. Κατόπιν, ως προς την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, συνεχίζεται η διακριτική μεταχείριση, γιατί λόγω του θέματος της μητρότητας είναι αιτία διακριτικής μεταχείρισης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάντως που δεχτήκατε να αναλάβετε αυτό το αξίωμα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κυρία Φιγκυρέιδο. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μπασελέ για να σχολιάσει όλες αυτές τις παρατηρήσεις και να δώσει απαντήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, όλους ε, τους βουλευτές ε, που σχολίασαν αυτά τα θέματα και έθεσαν ερωτήσεις. Ένα από τα θέματα είναι πώς συντονιζόμαστε με τις λοιπές υπηρεσίες και οργανισμούς των ΟΗΕ. Τι κάνουμε, μελέτη αντικτύπου. Δηλαδή, ξέρετε, Ένας από τους στόχου μας είναι κανονιστικός να θέσουμε τα βασικά πρότυπα. Κατόπιν υπάρχει και ένα επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή όλα τα προγράμματα και οι δράσεις που συνδέονται με αυτά τα θέματα, εφαρμογή των ψηφισμάτων, διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο κτλ. Τρίτο κομμάτι ε, είναι η λογοδοσία και ο συντονισμός. Ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε εάν ολόκληρο το σύστημα του ΟΗΕ λειτουργήσει καλύτερα, θα είναι προς όφελος ε, των γυναικών όλου του κόσμου. Έχουμε αναλάβει εντολή για να αναβαθμίσουμε το συντονισμό και εργαζόμαστε επ' αυτού, αλλά σημαντικό για μας είναι ε, η λογοδοσία. Δεν είμαστε αστυνομία για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά ε, θεωρούμε ότι δίνουμε μια γενικότερη κατεύθυνση ως προς τις βασικές προτεραιότητες για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε συνέργειες. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, αλλά όχι μόνο. Μπορούμε να ε, αυτά που κάνουμε να τα κάνουμε καλύτερα και σε συνεργασία με τους δε. Και η βασική πρόκληση για τις γυναίκες είναι να έχουν ειδικό βάρος οι γυναίκες και οι δράσεις να έχουν αποτέλεσμα αυτό στη ζωή των γυναικών. Υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων, όλοι είναι πολύ φιλόδοξοι και περιμένουν να κάνουμε εμεί θαύματα στη UN Women. Εντάξει, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά σε συνεργασία μαζί σα ε, μόνοι μα δεν μπορούμε. Δεν έχουμε του απαιτούμενου ε, πόρου. Έχουμε δηλαδή οικονομικού πόρου, αλλά θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερου για να καλύψουμε αυτέ τι μεγάλε προσδοκίε ε, που υπάρχουν από πλευρά των γυναικών. Για το ψήφισμα 1325 αναφερθήκατε πολύ σε αυτό. Πραγματικά είναι μία από την διάσταση ε, αντιμετώπισης των ενόπλων σειράξεων και κατάσταση μετά ε, από τις σειράξεις. Ε, συνεργάζομαι στην κυρία Βάλστρομ για την ειδική συντονίστρια, ειδική εκπρόσωπος για αυτά τα θέματα, αλλά δεν έχουμε θεσμική εκπροσώπηση σε όλες τις χώρες και τις είπαμε ότι θα τις δώσουμε πεζικό σε εισαγωγικά, τόσο ώστε επιτόπου να μπορεί να επιτελεί τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει, πιλωτικά προγράμματα για σύστημα έγκαιρα έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου, ε, εντελεχέστερη ανάλυση των φαινομένων βία, ε, Συνεργαζόμαστε επίσης για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις ε, γυναίκες, για την παραγραφή ως προς τους δράστες των αξιοπίνων πράξεων και ενίσχυση των γυναικείων οργανώσεων. Ε, στο, σε πολλές χώρες Αφρικής και ε, στο Κονγκό μεταξύ άλλων θα γίνουν εκλογές, ε, οπότε είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την παρουσία των γυναικών ως υποψήφιες αν το επιθυμούν, αλλά όχι μόνο διότι οι εκλογές είναι μια στιγμή όπου υπάρχει κίνδυνος για βία, βιασμό, ανασφάλεια γενικότερα για τις γυναίκες είναι μια επικίνδυνη περίοδος. Σχετικά με τον διαμεσολαβητικό ρόλο των γυναικών επίσης ε, και αναφέρομαι και στη δική σας ερώτηση για την κατάσταση στην ε, Παλαιστίνη και πώς μπορούν ε, δηλαδή να λειτουργήσουν η ειρηνευτική διαδικασία οι γυναίκες στην Παλαιστίνη. Έχουμε συγκεκριμένα ένα πρόγραμμα και Παλαιστίνης γυναίκες συνεργάζονται με τις γυναίκες στο Ισραήλ για να οικοδομήσουν ένα πιο ειρηνικό περιβάλλον, για να λειτουργήσουν διαμεσολαβητικά. Ε, όμως σε πολλά μέρη του κόσμου δεν ισχύει αυτό. Σε πολλές αφρικανικές χώρες ε, ε, όσοι μετήχαν στις ένοπλες σειράξεις ε, έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ε, δίπλα με αυτού που είχαν την πολιτική εξουσία αλλά δεν εκπροσωπούνται οι γυναίκες πάντως. Στον τομέα τη διαμεσολάβηση και των διαπραγματεύσεων επιδιώκουμε να αυξηθεί ο αριθμό τη γυναικεία εκπροσώπηση. Εμεί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ποιο θα είναι διαμεσολαβητής αλλά μπορούμε να προτείνουμε πολλέ υποψηφιότητε με προσόντα, με δεξιότητες. Δεν θέλω πάντως να να χρησιμοποιείται αυτό σε δικαιολογία γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες, έχουμε ένα εκατομμύριο δολάρια, τριετές πρόγραμμα θα συστήσουμε, να ενισχύσουμε δηλαδή την ικανότητα των γυναικών, να υποστηρίξουμε το ρόλο ε, των ανδρών ως διαμεσολαβητών γιατί και κάποιοι από αυτούς δεν γίνονται δεκτοί στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Και επίσης έχουμε και την υπηρεσία ε, διατήρησης της ειρήνης όπου προετοιμάζουμε μία ειδική μονάδα ταχείας παρέμβασης και εκεί θέλουν να συμμετάσχουν ε, γυναίκες ε, Έχουμε ένα επίσης ε, ε, αστυνομικό σώμα γυναικών και ένα τάγμα στο στρατό στην Ιγυρία όπου συμμετέχουν οι γυναίκες και όχι μόνο συμμετέχουν ε, στις παρελάσεις αλλά καταδεικνύουν την ισχύ τους κατέχοντας αυτές τις θέσεις και οι γυναίκες νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Όταν βλέπουν αυτές τις γυναίκες που είναι μες στην αστυνομία, στο στρατό, δηλαδή λειτουργούν ως σύμβολα και ως πρότυπα. Γι' αυτό είναι σημαντικό σημαντικό να μιλήσουμε για την χειραφέτηση. Οι γυναίκες, ε, κάποιες γυναίκες μπορούν να αναλάβουν ρόλο προτύπου και έτσι οι υπόλοιπε γυναίκες μπορούν να τις ακολουθήσουν. Θα δουν δεν υπάρχουν προσκόμματα, μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Και ε, έχω και μια πολύ ωραία ιστορία γιατί τα Άλμα χαλώνουν την πρώην πρόεδρο της Φιλανδίας. 9 ε, χρόνια ήταν στο ύπατο το αξίωμα και πήγε σε ένα βρεφικό σταθμό και ρώτησε τα παιδιά τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε ε, και ένα αγοράκι ε, όταν ερωτήθη θέλετε να γίνετε πρόεδρος. Μα στη χώρα μου δεν γίνονται άντρες πρόεδροι, απάντησε το αγοράκι, οι γυναίκες γίνονται. Βλέπετε λοιπόν πώς μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη νοοτροπία. Ε, έχοντας ε, ε, τις γυναίκες αυτούς τους ρόλους πρότυπα. Είναι δύσκολο οι γυναίκες να ε, έχουν παιδιά, να εργάζονται, να ακούγεται η φωνή τους. Ε, η χειραφέτηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το, αντιλαμβάνεστε, μου δώσατε τόσα παραδείγματα κι εσείς. Ε, στην Τασμανία, σε, χώρες, σε πολλές χώρες νοτιού της Σαχάρας, ποιο είναι το γεωργικό δυναμικό, οι γυναίκες φτάνουν και σε ποσοστό 80, 85% για την έγκυα όμως η διοκτησία μόνο 2%, 2 μόνο είναι γυναίκες. Ε, κάποιες δεν έχουν τη δυνατότητα να κληρονομήσουν. Δηλαδή πεθαίνει από AIDS ο, ο άντρα παραδείγματο χάρη και δεν μπορεί να κληρονομήσει η γυναίκα. Το παίρνει ο θείο, ο κουνιάδο, ο μπατζανάκη. Ένα άντρα, εν πάση περιπτώσει. Ε, πρόσβαση στην ε, πίστη, στην καταναλωτική και επιχειρηματική πίστη, ε, τροποποίηση της νομοθεσίας για να έχουν ισότιμα δικαιώματα οι γυναίκες. Η κυρία Μπάουερ μας μίλησε για την μητρική θνησιμότητα. Θα επανέλθουμε σε λεπτομέρειες. Είναι ένα ιατρικό ζήτημα και άρα μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Πάρα πολύ σημαντικό στα Ηνωμένα Έθνη σε κάποια διάσκεψη ε, ε, συντόνιζα ένα πάνελ για αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνουμε πολλά, μπορούμε να κάνουμε πολλά. χώρα χρειάζεται ανάλυση, διαφέρει η κατάσταση, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζουμε σε κάθε χώρα να ε, τη βοηθήσουμε να αναλύσει ποιο είναι το πρόβλημα. Παράδειγμα, όταν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Χιλή, υπήρχε ένα δίκτυο που συμμετείχε ε, η πρόεδρος της Τανζανίας, ο Στόλτμπεργκ και κάποιοι άλλοι και στην περιοχή μου ε, χρησιμοποίησαμε τους δείκτες γιατί έχουμε πολύ καλούς δείκτες στη Χίλη με την Παραγουάη, με τον Ισημερινό και με τη Βολιβία που είναι οι χώρες που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες συνεργαστήκαμε για να ταυτοποιήσουμε ακριβώς τα προβλήματα. Σε κάποια μέρη δεν είχαν ΜΕΕΣ, για παράδειγμα στην Τανζανία η πρόεδρος ε, ε, ε, ε, προχώρησε στην εκπαίδευση 5.000 μεών. Κάπου αλλού χρειάζονται μεταφορικά μέσα για να πάνε οι γυναίκες κάπου να γεννήσουν. Δηλαδή δεν είναι οι ίδιες οι ανάγκες παντού. Δυστυχώ δεν είναι δικός μου τομέα αυτό τη υγείας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε ειδικό πρόγραμμα, γιατί ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Και είναι απίστευτο αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Δεν έχω χρόνο. Θέλουν και άλλοι πολύ το λόγο. Θα μου δώσετε στη συνέχεια πάλι το λόγο να ξαναπαντήσω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Μπασελέ. Τώρα η Αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, η κυρία Νικολάη, θα πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μπασλέ, με μεγάλη χαρά σας βλέπω εδώ ενώπιον μας. Πρέπει να σας πω ότι στη δράση σας βρήκα την απάντηση σε αυτή την ερώτηση που πολύ συχνά προβληματίζει τους Αμερικανούς. Γιατί ο καλύτερος άνθρωπος για μια θέση ε, συχνά είναι γυναίκα. Έχετε κάνει πάρα πολλά ε, και σε νευραλγικά υπουργεία και στο Υπουργείο Αμήνης και ξέρετε και πώς να προσεγγίζετε τα θέματα ε, στη συνέχεια όταν διατελέσατε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες ε, ε, ζώνες πόλεμης ένοπλης σύραξης, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα ήθελα να καλωσορίσω τα πρόσφατα μέτρα που ελπίζω να αποδειχθούν αποτελεσματικά. Και είμαι βέβαιη ότι εσείς ε, θα το εξασφαλίσετε αυτό. Έχω μια ερώτηση. Ήμουν μέλος για έξι χρόνια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ίνστρου. Αυτού του οργανισμού του ερευνητικού, ε, ακούω ότι σκοπεύετε να τον διοργανώσετε. Με ποιο τρόπο? Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη των Επιτροπών. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε έκαστος ένα λεπτό και δυστυχώς πρέπει να είμαι αυστηρή γιατί δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Η κυρία Γκουμάη πρώτη. Ε, στα Ισπανικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω ε, και συνεχίζω στα Αγγλικά. Ως ε, Ουγγαρέζα χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεστε κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Είναι πολύ ωραία αυτά ε, και ωραία τα έγγραφα που ψηφίζουμε, αλλά χρειάζεται τώρα και αντίστοιχη οδηγία για να γίνει πράξη. Λέτε ότι οι γυναίκε είναι φορεί τη ανάπτυξη. Εγώ θα το πήγαινα παραπέρα και θα έλεγα ότι είναι φορεί τη αλλαγή. Κάποιο ε, έχει πει ότι όταν εκπαιδεύει έναν άντρα, εκπαιδεύει έναν άντρα. Όταν εκπαιδεύει μια γυναίκα, εκπαιδεύει την κοινωνία ολόκληρη, γιατί οι γυναίκε διαπαιδεύουν τα παιδιά του. Ε, χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ για το πρόγραμμα που αναφέρατε. Βεβαίω χρειάζεται και ένα gender budgeting ε, και στον προπολογισμό να λαμβάνονται υπόψη τα θέματα του φύλου και μάλιστα με τρόπο πολύ σοβαρό. Μια σύντομη ερώτηση λοιπόν. Είμαι πεπισμένη ότι με τη δική σας παρουσία ε, θα πάει πολύ καλά ο οργανισμός. Είστε για μας όλους πρότυπο εδώ εσείς. Και θα ήθελα να σας πω ε, ποια θα είναι η πρώτη σας προτεραιότητα. Να μας πείτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαφράνκα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω εδώ την παρουσία της κυρίας Μπασελέ, που είναι από μια χώρα πάρα πολύ αγαπημένη για μας, τη Χιλή, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε να αναλαμβάνετε τόσο υψηλά καθήκοντα στα Ηνωμένα Έθνη. Το σχέδιο δράσεών σας είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και το έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή Εξωτερικών, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη και πιο συγκεκριμένα στη Γενική Συνέλευση, όπου έχουμε κάποιες δυσκολίες. Εδώ θα ήθελα να σας πω και κύριε Μπασελέ και στις προτεραιότητες που μας παρουσιάσατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιοι είναι οι πόροι, οι δημοσιονομικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που έχετε στη διάθεσή σας για να προχωρήσετε στους στόχους σας και πιστεύετε ότι θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπαριθμόν ένα χρηματοδότης ε, του ΟΗΕ στους διάφορους οργανισμούς μήπως θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πολιετές συμφωνό πλαίσιο, μια συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε ότι εδώ είμαστε στο πλευρό σας, ε, κυρία Μπασελέ, βρίσκεται πάντα πρόσφορο έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Σαλαφράγκα. Η κυρία Πλάμ τώρα. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ε, ε, καλωσορίσω εγκάρδια την κυρία Μπασελέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πρέπει να σας πω ότι ήμουν ε, εισηγήτρια για ένα σημαντικό θέμα που είναι το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, αυτό όμως είναι και διεθνές πρόβλημα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στόχος όλων μας είναι η καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών. Μια που είστε και γιατρός και ταυτόχρονα μία από τις πιο ισχυρές πλέον γυναίκες στον κόσμο και ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή τη θέση που αναλάβατε ε, τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τη μελλοντική μας συνεργασία ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό φαινόμενο της φτώχειας των γυναικών. Γιατί η φτώχεια είναι όντως γένους θηλυκού και η μετανάστευση είναι γένους θηλυκού και θα πρέπει από κοινού να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σημαντικά φαινόμενα. Ένα τελευταίο, Πρόεδρε, και κλείνω. Τον Ιούνιο φέτος θα καταθέσετε στο εκτελεστικό συμβούλιο το στρατηγικό σας σχέδιο. Μπορείτε να μας δώσετε ήδη κάποιες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ένστ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι κυρία Μπασλέ που είστε στο Κοινοβούλιο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Μια ερώτηση έχω πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ο λεγόμενο όρο και ρύθμιση του 30%. Στη Γερμανία αυτό το περίφημο 30% έχει καταρρεύσει. Γιατί έβαλε βέτο μία καγκελάριος, γυναίκα κατά τα άλλα, η κυρία Μέρκελ, που είπε ότι δεν επιτρέπεται νομοθετική ρύθμιση, δεν μπορεί να επιβάλλεται αυτό δια νόμου, να είναι εθελοντικό και τέρμα η συζήτηση. Στη Γερμανία, στη δικαιοσύνη ας πούμε, είναι ένας χώρος ελεύθερος γυναικών θα μπορούσαμε να το πούμε. Σχεδόν καμία γυναικεία παρουσία ε, στους δικαστές και στη λήψη των αποφάσεων. Και σε άλλους τομείς ισχύει αυτό. Και στην οικονομία σε μεγάλο βαθμό είναι καταστροφή για μια τόσο πλούσια χώρα και με τόσο δημοκρατική. Και σας ερωτώ λοιπόν, είπατε ότι πέντε είναι οι χώρες που επέβαλαν ε, χωρίς νομοθεσία αυτό το 30% συμμετοχή των γυναικών. Πώς τα κατάφεραν χωρίς νομοθεσία. Και στις υπόλοιπες τι γίνεται. και που υπάρχει νομοθεσία πώς επευλήθη και υλοποιήθηκε στην πράξη. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μουνής. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Μπασαλέ, που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη σας επίσκεψη στις Βρυξέλλες και μάλιστα τέτοιες στιγμές που πιστεύω ότι τα μεγάλα διεθνή γεγονότα δεν μπορούν να επισκιάσουν ε, ε, αυτό το σημαντικό θέμα του mainstreaming και της ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των γυναικών. Στις 7 Μαου του 2009 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για την ένταξη της διάσταση του φύλου σε εξωτερικές σχέσεις ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα τα τη διάρκεια τη ζωή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι άπειρα τα ψηφίσματα για την ισότητα, για την ίση αμοιβή των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τι γενικέ δηλώσει όμω, αυτέ τι γενικέ θέσει, όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσουμε συγκεκριμένα μέτρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένε πολιτικές ομάδες δεν είναι τόσο σαφείς. Για ποσοστώσει μιλάω ή για την ε, ε, αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία των γυναικών. Και στις χώρες μας το ίδιο. Ε, η σοσιαλιστική κυβέρνηση σαν πρώτο νόμο πέρασε ε, ε, το νόμο κατά της βίας με βάση το φύλλο. Και πολλοί λένε ωραία λόγια και μεγαλόστομα, αλλά όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσουν δεν τα κάνουν αυτά πράξη άλλα κόμματα. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η δική μου δέσμευση. Ως συγγήτρια για τον προπολογισμό του 2012 στην Επιτροπή Εξωτερικών και για τους διεθνείς οργανισμούς τους πολυμερείς θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, είναι μεγαλύτερη στα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, να διοχετεύονται συγκεκριμένα κονδύλια, τουλάχιστον σε κάποιο ποσοστό, ε, προς ε, τη δική σας οργάνωση, ο ΙΕ Γυναίκες. Ερώτηση τώρα πώς εξασφαλίζεται ο εγκάρσιος χαρακτήρας και η συνεργασία με τους άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ. Um, και προσπαθείτε να τηρήσετε το χρόνο σας. Θα προσπαθήσω και θα μιλήσω στα ισπανικά. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά που αισθάνομαι που σας βλέπω εδώ όχι μόνο λόγω της προσωπικής σας και πολιτικής ιστορίας και ζωής που ανάφεραν και άλλοι, αλλά και για το όραμα που μας δίνετε και αυτό που θέλετε ε, ως γυναίκα να επιτύχετε. Και συνεχίζω στα αγγλικά. Χάρηκα πάρα πολύ ε, που μας είπατε για το όραμά σας, για τις γυναίκες και τους άνδρες στην κοινωνία μας. Θα πρέπει ε, να ε, δούμε ότι ε, είναι πολλά τα εμπόδια και οι γυναίκες χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες για να τα πετύχουν. Θέλω να σας ρωτήσω τρία θέματα. Πρώτο, τι προϋπολογισμό έχετε ε, στην οργάνωση του ΟΗ για τις γυναίκες. Γνωρίζω ότι στο παρελθόν ήταν μόνο εθελοντικές οι συμμετοχές των κρατών. Έχει αλλάξει αυτό στα Ηνωμένα Έθνη, είναι υποχρεωτική. Μιλήσατε για το ψήφισμα 1325, υπάρχει και άλλο το 1820 για τη βία κατά των γυναικών τη σεξουαλική ε, σε πολέμους και στο Κονγκό. Το είπε η Εύα Ζολή, ε, υπάρχει καμία προσπάθεια για πρόληψη αυτό. Και το τέλος, ε, τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση, αντισύλληψη ή τα δικαιώματα των λεσβιών ε, να πούμε ότι μια γυναίκα δεν είναι ε, απαραίτητο να παντρευτεί για να ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσε. Κυρία Ρομέρα, έχει τώρα το λόγο. Καλώς ορίσατε κυρία Βασιλέ. Και εγώ στα Ισπανικά, Ισπανίδα είμαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς για τη βία κατά των γυναικών, διότι είπατε ότι σε πολλές χώρες δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δεν έχει φτάσει πλέον η ώρα να υπάρξει σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Και εσείς να δώσετε την όθηση από τη σημερινή σας θέση, έτσι ώστε να οριστεί αδίκημα αυτό η βία κατά των γυναικών σε όλες τις χώρες και να συμπεριληφθεί στον ποινικό κώδικα και να μην είναι πλημέλημα, αλλά είναι κακούργημα. Σε πολλές χώρες δεν θεωρείται κακούργημα και αφήστε δε που είναι ταμπού. Και όταν είναι ταμπού είναι ένα δίκημα ποινικό το οποίο δεν μπορεί να διωχθεί εάν αποσιωπάται και δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης γίνεται η προσπάθεια, θα προτείνουν μια σύμβαση ε, ε, κατά τη βίας η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να κάνει οδηγία. Εάν αυτό συνέπιπτε και με μια σύμβαση του ΟΗΕ σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαμε να εντείνουμε την πρόληψη και να έχουμε και αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων. Για να μην είναι μόνο ένα θέμα πρόληψης με ε, διαταγές ε, προστασίας στην Ευρώπη, αλλά διεθνές. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρομέρο. Η κυρία Μπιλμπάο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μπατσελέτ που ήρθατε. Έχω έρθει στη Χιλή ως πρόεδρος του Βασκικού Κοινοβουλίου ε, στην αρχή ε, της προεδρίας σας κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας τότε και θυμάμαι τα αρχικά μέσα που λάβατε και τα μέτρα τα κοινωνικά που ε, ε σας επιτέθηκαν πολύ με επικρίσεις και σήμερα κανείς δεν τολμάει ε, όχι να τα αποσύρει ούτε να τα επικρίνει. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη δράση σας στη χώρα σας. Βεβαίως οι γυναίκες εμείς εργαζόμαστε, βοηθάμε στην ειρήνευση, ε, στην εκπαίδευση, στην ανατροφή των παιδιών. Οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι πιο ανταγωνιστικές, ε, αγωνιζόμαστε παντού αλλά στην πολιτική απουσιάζουμε. Αναφέρατε κάποια στοιχεία Όπου πετύχαμε το κάναμε ακριβώς λόγω μηχανισμών. Και το κοινοβούλιο εδώ ε, δεν είναι ομόφανο όμως αυτά. Υπάρχουν ακόμα αντιστάσεις. Γι' αυτό χρειάζονται πολιτικές ε, θετικής δράσης. Υπάρχει μεγάλη αντίσταση ανδρική, ε, οι οποίοι σαστίζουν όταν βλέπουν τις γυναίκες στην πολιτική. Στις πολιτικές που αναφέρατε, έχετε σκεφτεί να καταπολεμήσετε τα στερεότυπα, δηλαδή το ανδρικό πρότυπο, τελειώνω, ε, να μην είναι το παλιό ανδρικό στερεότυπο, υπάρχουν νέες μορφές ανδρών. Πρέπει να προβάλλουμε τη σημερινή εικόνα του άνδρα, όχι το στερεότυπο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κώστα τώρα. Είμαι ευτυχή που σα γνωρίζω άμεσα. Πολλοί από εμά σα παρακολουθήσαμε την πορεία σα ακόμα και από μακριά και εμεί στη χώρα μα ε, ε, στην Ιταλία. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να ρωτήσω σε σχέση με τα πολλά που ήδη υπόθηκαν ε, να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ένδυας που όντως έχει γυναικείο πρόσωπο και παιδικό πρόσωπο ε, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που να μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο της δικής σας γραμματείας και πιο συγκεκριμένα εμείς εγκρίναμε στο Ευρωκοινοβούλιο μετά από το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ένδυα ε, δουλεύουμε για μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της στόχες και μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις ε, που αναλάβαμε είναι μια πρωτοβουλία για τις μικροπιστώσεις και μικροχρηματοδότηση. Πέρα από τις συζητήσεις που γίνονται σε διεθνές επίπεδο, θα ήθελα να καταλάβω αν εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια ισχυρή πρωτοβουλία, γιατί στόχοι είναι οι γυναίκες, η αυτονομία τους και το κατόφλι φτώχειας. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά τη σχέση ανάμεσα στη δική σας γραμματεία και την Επίτροπη Ελέγχου των Διακρίσεων. Ε, ε, είναι δύο διαφορετικοί οργανισμοί, υπάρχει όμως τρόπος επικοινωνίας για την νομίζω πως υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα στις δύο ε, πρωτοβουλίες αυτές. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστούμε κυρία Κώστα. Υπολείπονται κάποιοι ομιλητές. Πραγματικά δεν μπορείτε να υπερβείτε το ένα λεπτό, αλλιώ ε, δεν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε την κυρία Μπασελέ γιατί θα αποχωρήσει στις 10.30 η κυρία Κράτσα τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Μπασλέ, ε, έχετε ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχει ταύτιση των απόψεων και των στόχων που υπηρετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά των αξιών για την ε, ε, ισότητα ανδρών και γυναικών, για την κοινωνία δικαιοσύνης χωρίς διακρίσεις και για τη δημιουργία ενός κόσμου με δικαιοσύνη και ειρήνη που αποτελούν ως προϋπόθεση την ισότητα. Ε, Πιστεύω λοιπόν ότι η συνεργασία μας μπορεί να είναι πολύ επικοδομητική. Αυτό που μένει σήμερα και πιστεύω θα, η επίσκεψή σας θα σηματοδοτήσει κάτι σημαντικό είναι να θέσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Η ανταλλαγή απόψεων, η επικοινωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και των ε, υπηρεσιών σας θα είναι πολύ σημαντικές για να επικαιροποιούμε πάντα τους στόχους μας και τους μεθόδους μας αλλά είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, να αποτελέσει επίσκεψή σας την αρχή ενός, τη, τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε κυρία Κλάς τώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Μπασελέκα, σα ορίσατε στην Ευρώπη. Εγώ είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω με την Επιτροπή, την Αντιπροσωπεία της Χίλης ως πρόεδρο της χώρας σας, πάρα πολύ δυναμική ε, και σπουδαία και χαίρομαι που αναλαμβάνετε τώρα αυτά τα καθήκοντα και στο πρόσωπό σας πραγματικά Έχουμε πολλές ελπίδες. Είπατε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε και τους άντρες, γιατί από κοινού θα πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε έχω την ερώτηση, έχετε ένα προϋπολογισμό να διαχειριστείτε, ωραία, αλλά όσο έχετε πρόσβαση και σε άλλα πράγματα και οικονομικά. Και εγώ που είμαι η συγκήτρια για το νερό στην ΑΚΕ, οι γυναίκες παίζουν πάρα πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Και ήθελα ε, να πω ότι είναι αλληλένδετο όλα αυτά και εγκάρσιες οι πολιτικές και αγωνιζόμαστε για τις γυναίκες παντού. Αναφέρατε τις εκλογές στο Κονγκό και θέλετε να καλέσετε τις γυναίκες να πάνε να ψηφίσουν. Μα είναι το εκλογικό δίκαιο στο Κονγκό τόσο αντιδημοκρατικό που δεν πρόκειται να είναι δημοκρατικές εκλογές ούτε για τους άνδρες ούτε για τις γυναίκες. Κοιτάξτε και αυτό το θέμα σας παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόμες είναι η τελευταία ομιλήτρια. Πρόεδρε, στα τέλη της εβδομάδας ε, θα συναντηθούμε στο Κάιρο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας σχετικά με αυτά που μπορούμε να κάνουμε στη Βόρεια Αφρική και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο για τις γυναίκες ε, γιατί είναι στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη μεταβατική περίοδο προς τη δημοκρατία οι γυναίκες. Ήρθα σε επαφή με γυναίκες στην Αίγυπτο και εσείς το ίδιο φαντάζομαι. Και έπαθα σοκ γιατί στην ε, πλατεία τα χρήστη ε, ε, και μετά σε άλλα μέρη ε, υπέστησαν ε, επιθέσεις, οι γυναίκες ε, Σε έκαναν υποχρεωτικά επίσης ε, τεστ ε, Παρθενία αν είναι δυνατόν. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τα συμπεράσματά σας. Mrs. Κυρία Τόμψεν. Thank you, Σας ευχαριστούμε, κυρία Μπασελέ, που ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κάτι για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ε, πέρσι είχαμε μία εκστρατεία με τίτλο ε, «Σώμα μου είναι, άρα έχω δικαιώματα επ' αυτού». Ε, Ήταν μία καμπάνια των σοσιαλιστών και Βλέπουμε ότι παρά τα αποτελέσματα που έχουμε ήδη, έχουμε ακόμη προβλήματα για τη μητρική εθνισμότητα. Υπάρχει πρόβλημα διότι, να σα εξηγήσω, χτες ε, συζητούσαμε με Παλαιστίνιες γυναίκες και έχουν το υψηλότερο ε, επίπεδο γεννητικότητας στον κόσμο. 10 μέχρι 10 παιδιά κάνουν και καταλαβαίνετε, γιατί και εμείς ε, γυναίκες είμαστε, δεν θέλουμε συνέχεια να κάνουμε παιδιά. Ε, γι' αυτό και φίβραμε την αντισύλληψη, πολλούς τρόπους αντισύλληψης ε, θεωρώ ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός πρέπει να είναι στην καρδιά των προβληματισμών μας. Ε, ευχαριστούμε και η κυρία Κράτσα θέλει να κάνει σύντομο σχόλιο, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο, ήθελα να πω κάτι το οποίο θεωρώ σημαντική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε προηγουμένως η προσπάθεια για την συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και αναφέρθηκαμε στα πρότυπο της Νορβηγίας, τώρα μπορούμε να είμαστε ε, ευχαριστημένοι και περήφανοι και για τις κατακτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη υπάρχει νόμος σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο, στις κάτω χώρες. Η συζήτηση είναι πολύ συγκεκριμένη προς αυτή την κατεύθυνση στην Ιταλία, στο Βέλγιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει υπό επεξεργασία μια έκθεση που έχω την τιμή να είμαι εισηγήτρια και ίσως γνωρίζετε και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουμε σε νομοθετική κατοχύρωση εάν οι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων δεν καταλήξουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κράτσα και θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μπασελέ. Πάρα πολλά ερωτήματα έχετε να απαντήσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς έχω λιγότερο από ένα λεπτό. Ε, πιθανότατα δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα αλλά όπως σας είπα είναι οι αρχές μιας σχέσης. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί πιστεύω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ερωτήσεις δηλαδή πώς μπορούμε από κοινού να τα καταφέρουμε, να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας, να σταματήσουμε παράλληλα να κάνουμε πράγματα που μπορεί να είναι πολύ σημαντικά μεμονωμένα, αλλά να μην έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη βελτίωση της ζωής των γυναικών. Και όσον αφορά τις ευκαιρίες, το Ντέρμπαν, το Ρίο για παράδειγμα, Ρίο συν βιώσιμη ανάπτυξη και εκεί πρώτη φορά μάλιστα στην Κανκούν αναφέρθηκε κάτι για τις γυναίκες και τις κλιματικές αλλαγές. Ήμουνα τόσο πεπισμένη ότι είναι σημαντικό ο αντίκτυπο. Οι γυναίκε δέχονται διαφορετικό αντίκτυπο, αλλά είναι και μέρο τη λύση. Δουλεύουμε γι' αυτό, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν έχαμε πολλή εμπειρία μέχρι στιγμή όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες στο προσωπικό μας, αλλά θα συνεργαστούμε με ΜΚΟ, με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στον τέρμπον και στο Ρίο Συνήκωση θα έχουμε ένα σημαντικό μήνυμα για τις... Ε, για τους στόχου τη χιλιετία ε, είναι παράδοξο. Είναι ένα από τα θέματα και τι προκλήσεις που έχουμε να κάνουμε. Ε, πολλά λόγια Ακούμε ε, ωραία λόγια για τις γυναίκες, αλλά επιτεύγματα δεν υπάρχουν αρκετά. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε ακόμα να κάνουμε. Και κάτι για το οποίο εργάζομαι είναι ότι είμαι πεπισμένος πως τα δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά βέβαια για αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων δεν είναι αυτό το καλύτερο επιχείρημα. Για περιμένουν να αλλάξουν στάση, να ρίσουν τον προπολογισμό και αυτά είναι πιο σημαντικά. Όσον αφορά λοιπόν τις πολιτικές και κοινωνικές υποθέσεις, ε, αυτό το να συνεχίζουμε με την Ίνστρο θα είναι ένα κέντρο κατάρτισης αλλά θα φέρουμε στο Γενικό Επιτελείο τη λειτουργία της έρευνας. Όχι για να κάνουμε εμείς την έρευνα αλλά για να φτιάξουμε ένα μεγάλο δίκτυο με τα πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο, με κέντρα αριστείας, με κέντρα έρευνας τα οποία ήδη ε, κάνουν πολλά ώστε εμείς να χρησιμεύσουμε σε ένα χρηματιστήριο γνώσης, να διαδώσουμε παντού τις γνώσεις αυτές για να αποδείξουμε πόσα χάνει ο κόσμος χωρίς να δίνει, επειδή μάλλον δεν δίνει ευκαιρίες στις γυναίκες. Θέσατε μια πολύ σημαντική ερώτηση, κυρία Στρέλα, για την συμφιλίωση της πολιτικής ζωής με την ε, προσωπική ζωή. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας δώσω πολιτικό ορθή απάντηση. Πολιτικό ορθό, θα, θα, σαν ήθελα να μιλήσω, ε, είναι να πω ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να κάνουμε κάτι μπορούμε. Αλλά αν θέλω να μιλήσω ειλικρινά θα πρέπει να σας πω ότι, δεν είναι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει μια απλή γυναίκα. Θα απλή, η γυναίκα μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά όχι όλα ταυτόχρονα. Και όταν μπορείς να τα μάθεις αυτά, ίσως να αισθανθείς λιγότερο ένοχη. Γιατί όλες μας θέλουμε να είμαστε υπεύθυνε. Να είμαστε υπεύθυνε, να είμαστε τέλειες, να έχουμε ένα ωραίο σπίτι. Τα παιδιά μας να είναι ευχαριστημένοι Μα τα παιδιά ποτέ δεν είναι ευχαριστημένα όταν δουλεύουμε πολύ ή όποια και αν είναι η δουλειά μας αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε κάτι Δηλαδή να αλλάξουμε την ποσότητα με ποιότητα. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί ποτέ να είναι και πολύ, πολύ επιτυχημένο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι κι αλλιώς και είναι αυτό κομμάτι της ζωής. Προχωράνε οι γυναίκες σε πάρα πολλούς τομείς, οπότε σε λίγο δεν θα είναι ευθύνη μόνο της γυναίκας να έχει ένα υπέροχο σπίτι, υπέροχα παιδιά πανευτυχή, θα είναι ευθύνη όλες τις οικογένειες. Και τι να κάνεις, να κάνεις, ε, να πας τα παιδιά στον ψυχολόγο, όταν ήμουν πρόεδρος, ναι, για να σκεφτούμε α, γιατί εγώ να είμαι διαφορετική από έναν άνδρα πρόεδρο ας πούμε ας πούμε για τα παιδιά το, μάλλον και ένας άνδρας πρόεδρος το ίδιο απόν εγώ ήμουν και μόνη είχα τη μητέρα μου που με βοηθούσε ευτυχώς αλλά πάντως απάντηση εύκολη δεν υπάρχει αν ανοίξουμε δρόμους και παράθυρα για ευκαιρίες και αν περισσότερες γυναίκες ασχολούνται με την πολιτική και τις διάφορες, τα διάφορα πόστα θα βρούμε τρόπους, θα αναπτύξουμε περισσότερους παιδικούς σταθμούς, βρεφονιπιακούς σταθμούς, θα διευκολύνουμε τη ζωή των γυναικών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα σωρό θέσεις και δουλειές. Αλλά σαφώς ο συνδυασμός της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή είναι κάτι που θα πρέπει να το πετωπίσουν και οι επιχειρήσεις, πώς θα διευκολύνουν τους γυναίκες υπαλλήλους από τις οικογένειες και από τους συζύγους, τους ε, άνδρες όταν υπάρχουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κάτι να πω δύο λόγια για την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντική ως σύμβολο. Συζητούσα με νέα κορίτσια, δεν ξέρω να σας το ανέφερα, την, την, την, την γενιά του Facebook όπως λέγεται και τη γενιά του Twitter. Αυτό ήταν πολύ ωραίο γιατί ενώ συνομιλούσαμε ήταν με τους υπολογιστές τους και ε, ε, χτυπούσαν τα όσα λέγαμε. Πολλοί δηλαδή συμμετείχαν ε, στην συνεδρίαση ακόμα και αν δεν ήταν, απόν, δεν ήταν παρόντες. Ήμασταν εκεί, αλλά τώρα όχι. Είμαστε αόρατοι. Πήγαμε εκεί και μας είπαν, κοιτάξτε, πρέπει να είστε λογικοί, είναι πολύ ασταθής η κατάσταση, πρέπει να περιμένετε. Αφήστε να εδραιωθεί η κατάσταση, να σταθεροποιηθεί και μετά θα ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εγώ τις είπα τις ιστορίες από όλα τα μέρη όπου οι γυναίκες φάνηκαν λογικές, ακόμα περιμένουν. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Γιατί οι πολιτικές εξελίξεις όντως δεν είναι σαφείς, τα, νέα κόμματα είναι αδύναμα, δεν ξέρουν πώς θα τα πάνε στις εκλογές και στις κοινοβουλευτικές και τις προεδρικές. Εγώ νομίζω μπορούμε να κάνουμε πολλά. Τι χρειάζεται υποστήριξη. Χρειάζονται υποστήριξη, πείρα, Αυτά τα κορίτσια είπαν «Ε, θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τα κάνουμε. Ποτέ δεν έχουμε φτιάξει, στήσει μια οργάνωση, δεν ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε. Όταν θα πάω πίσω στη Νέα Υόρκη θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για να στηρίξουμε αυτές τις οργανώσεις νέων που είναι σπουδαίες, είναι καταπληκτικά έξυπνοι και ενθουσιώδεις αλλά και οι πιο ηλικιωμένε γυναίκες μπορούν να είναι ε, ευφυεί, υπέροχε ε, και να καταφέρουν πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να το στηρίξουμε ε, να φτιάξουν ένα Υπουργείο για τα θέματα των φίλων, όχι ότι θα τους φτιάξει αυτό αυτόματα ισότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει στο ε, Υπουργικό Συμβούλιο κάτι μπορεί να κάνουν. Και έπειτα με το mainstreaming υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα όταν ε, θες να κάνεις main, mainstreaming στην ατζέντα, γιατί όταν κάτι υποτίθεται είναι παντού τελικά καταλήγει να μην είναι πουθενά. Ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στον προπολογισμό και αλλού παντού θα ε, αναφέρεται σαφώς το θέμα των φύλων. Όταν είναι στο mainstream πολύ συχνά ξεχνιέται. Καλό είναι να μπαίνει στο mainstream, αλλά καλύτερα είναι να είναι πιο συγκεκριμένο. Τώρα, πληθυσμός, ε, αναπορικά δικαιώματα κτλ. Πρέπει να σκεφτούμε παγκόσμια στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Το 2050 αν ναι, ε, το 2050 θα είμαστε 9 με 10 δις πάνω στην γη. Αλλά οι χώρες που αυξάνουν τα ποσοστά γεννητικότητας είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες. Και επίσης, ε, ζούμε περισσότερα χρόνια και Έχουμε πολλές χρόνιες ασθένειες, όχι μεταδοτικές. Να τα πούμε πιο απλά, θα είμαστε περισσότερο, περισσότεροι, ε, όχι πιο πλούσιοι και με χειρότερη υγεία. Περισσότερη φτώχεια θα υπάρχει, δηλαδή έλλειψη ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Να, πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν τους πληθυσμού. πρέπει να σκεφτούμε τον οικογενειακό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Είναι κάτι αυτό αλλά όταν δουλεύουμε με το UNPA ε, πρέπει να συνδυάσουμε και τις υπηρεσίες εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν δίνεται μεγάλη προσοχή, αρκετή προσοχή σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να ασχολούμαστε καθυστερημένα με όλα τα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε λύσεις να προλάβουμε τις πρόερες εγκυμοσύνες, τις πρόορους γάμους, τις βιασμούς, ένα σωρό πράγματα, την μόλυνση με, με το AIDS, να βρεθεί θεραπεία και η, γυναίκα να μην ε, ε βοηθάτε μόνο όταν ε, είναι έγκυος και θα κάνει παιδί, αλλά και μετά να μπορέσει να επιβιώσει. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε μαζί. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Νομίζω πως υπάρχουν ένα σώρο πράγματα που πρέπει να κάνουμε, οι γυναίκες και οι άνδρες και προσπαθούμε να κάνουμε συμμαχίες με τους άνδρες για όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς και πολλούς ακόμη. Έχουμε πολύ σπουδαίους πρωταθλητές, αλλά χρειαζόμαστε πολλούς περισσότερους είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθω να έχουμε ισότητα φίλων και σε αυτή την αίθουσα. Όχι μόνο γυναίκες πολλές, αλλά και πολλούς άνδρες να έχουμε θα είναι πολύ καλύτερο να μην χρειαζόμαστε επιτροπή γυναικών ε, πια. Ε, όταν τη ρωτήσαμε, ναι, ναι χρειάζεται την Έλληνα Ρούσβελ, δεν χρειάζεται ειδική επιτροπή για τις γυναίκες, ε, είπε τότε ναι, αλλά και μετά από 60 χρόνια εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε αυτή την επιτροπή. Βασίζομαι λοιπόν σε εσά και στη συνεργασία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπασελέ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Βλέπουμε τις εμπειρίες σας, την αφοσίωση που δείχνετε, τη βούλησή σας να προχωρήσετε